Πιμέντα Λόπες, της κυρίας Καρολίνα Πουνσέτ Μπανέλ και του κυρίου Γιάρο Μυρκόλτσερ και πρότεινε <clears throat> με ε, ημερομηνία 31η Ιανουαρίου 2016, 3 Φεβρουαρίου και 4 Φεβρουαρίου να θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί η εντολή του. Υπάρχουν αντιρρήσει. Επομένω, οι εντολέ αυτέ έχουν επιβεβαιωθεί. Η κυρία Φον Στόρχ έχει φύγει από την